Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο. Κοιτάξτε, δεν με πειράζει αν ε, μου είπα να το βουλώσω. Όπως μου είπε ο αξιότιμος ε, κύριος του Γιούκη που μας έκανε μάθημα για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όταν όμως έρχεται άλλος και με αποκαλεί φασίστα, νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το όριο. Ε, το συγγνώμη γιατί δεν γνωρίζω όλα τα μέλη του UKIP ε, με τα μικρά τους ονόματα, όμως περιμένω μια συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Miss you have the floor. Mi ε, ε, λυπάμαι για αυτή την προσβολή που μας απευθύνατε. Ε, την έχουμε δεχτεί πάρα πολλές φορές, την ε, κατηγορία την πασιαφασίστη. Σας είπα προηγουμένως ότι εμάς, μας αδειάζει η κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι προσβολή. Θέλω να επανέλθω όμως στο θέμα του κανονισμού. Το άρθρο 191 λέει ότι σε περίπτωση που αναστέλλεται μία συζήτηση η ψηφοφορία θα πρέπει να λάβει χώρα άμεσα και όχι μετά από διακοπή 30 λεπτών. Έτσι κι και αυτό δεν έχει σημασία. Γιατί ο δικό μα ο στόχο δεν ήταν να διακόψουμε τη συνεδρίαση. Μα ενδιέφερε πάρα πολύ το ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπω είναι το Μπουρούντι και εμεί είμαστε πεπισμένοι για τη σημασία αυτού του θέματο, ήταν παρόντε το πολύ 5 ή 6 άτομα για συζήτηση. Είμαι όμω χαρούμενη για το γεγονό ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα, δηλαδή το να ισχύει ο κανισμό, αλλά Όποτε σας αρέσει εσάς, τότε ήρθατε όλοι. Να ειδού. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ το αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ενημερώσω τους βουλευτές και τις βουλευτές ότι πράγματι αυτό συνέβη βάσει του άρθρου 191. Έχετε άλλο διαδικαστικό θέμα να θέσετε κυρία μου παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά κοιτάξτε, ούτε κι εγώ ούτε και οι συνάδελφοί μου θέλουμε να αφήσουμε απαρατήρητη τη μεγάλη προσβολή που μας απευθύνατε, που απευθύνεται και σε εμά ότι είμαστε φασίστες. Είναι απαράδεκτο αυτό εκ μέρου ενός συναδέλφου. Αυτό αποτελεί κατάφορη παραβίαση του κανονισμού, άρθρο 11, κατάφορη παραβίαση της ε, έκφρασης, ελευθερίας έκφρασης. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κατηγορεί κάποιον ως φασίστα, κυρίως εκείνοι οι οποίοι έχουν και αυτή ευθύνη ε, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κυρίως για το ότι είχαν εγκλειστεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης οι μαχητές. Σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας. Παρακαλώ για την υπομονή και την επίοικιά σας. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Ζητώ από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιδεικνύουν υπομονή, να ακούν ο ένας τον άλλον και να ακούν και εμένα όταν παίρνω το λόγο για να σας πω τι συνέβη στην αίθουσα της Ολομέλειας. Μπορεί να υπάρχουν μέλη που να ενδιαφέρονται λοιπόν. Και γι' αυτό λέω ότι σε σχέση με το ε, άρθρο 191 επί θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Eh, Μια συγκεκριμένη ερώτηση διαδικαστική και πολύ σημαντική για μένα. Παρόλο που αλλάζω λίγο το θέμα. Βλέπω ότι η κυρία Γιούτο βρίσκεται εδώ μαζί με το μωρό τη. Ο κύριο Σούλτ από την άλλη μεριά μου είχε απαγορεύσει να μπω σε αυτήν την αίθουσα με την κόρη μου 8 μηνών. Γιατί αυτή η διάκριση. mégiscsak folytatnánk ezt az ülést ε, προτείνω να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Βάσει λοιπόν του κανόνα 191, η πολιτική ομάδα EFTD ζήτησε να διακοπεί η συνεδρίαση. Θέλετε να διατηρήσετε το αίτημα που έχετε υποβάλει. Στρέφουμε προς το EFTD. Εάν ναι, θα τεθεί προς πληροφορία το αίτημά σας. Επομένως, τα μέλη που ζητήσατε τη διακοπή της συνεδρίασης. Όποιοι είναι υπέρ. Κύριε Γούλφ, θέλετε το λόγο. Okay. You don't want the vote to happen. Okay. Mad Can you hear me, Madam Chairman? Με ακούτε, κυρία Πρόεδρε. Γιατί δεν φαίνεται να λειτουργεί το μικρόφωνο μου και δεν είμαι σίγουρος. Με ακούτε, καλώς. Θέλετε οι υπόλοιποι να ακούσετε αυτό που έχω να πω ή όχι. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να στέκομαι όρθιος για όση ώρα χρειαστεί μέχρι ότου μου πείτε ότι με, ότι με ακούτε γιατί θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας. Έχετε δίκιο. Βάσει του 191 υποβάλαμε αυτό το αίτημα στην αίθουσα της Ολομέλειας όταν ήταν άδεια. Ελπίζω να πρόλαβαν να απολαύσουν το ποτό τους μέχρι που ήρθε το μήνυμα του Twitter και το email να τους διακόψει από τα ε, πάρα που έπιναν το ποτό τους στο κτίριο και να έρθουν στην Ολομέλεια οι υπόλοιποι. Συγγνώμη κύριε, θέλετε να πάρετε το λόγο και να μιλήσετε εξ ονόματός μου. Ε, ευχαρίστω σταματάω να μιλάω από τη στιγμή που με διακόπτετε. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο, αν θέλετε, υποχωρώ. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Πρόεδρε, ε, σας ε, διατυπώσαμε το κανόνα με απόλυτη σαφήνεια, γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Και λέει ο κανόνας 191 ότι μπορεί να διακοπεί μια συνεδρίαση κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Και ήμασταν σε συζήτηση. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει κάτι τέτοιο κατόπιν πρότασης του Προέδρου ή αιτήματο πολιτικής ομάδας. Και εμείς υποβάλαμε τέτοιο αίτημα ως πολιτική ομάδα. Τέτοια πρόταση θα ε, τεθεί προς πληροφορία αμέσως. Αυτό ζητήσαμε. Όμως η ψηφοφορία ανεστάλει, διακόπη για 30 λεπτά. Μετατέθηκε 30 λεπτά αργότερα. Τώρα δηλαδή. Επομένως, η πολιτική ομάδα αποχωρεί για να σκεφτεί τις επόμενες δύο ώρες κατά πόσο ε, θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να επανέλθουμε και να υποβάλουμε εκ νέου τέτοιου είδους αίτημα. Θα εξετάσουμε τις ε, νομικές ε, συνέπειες, θα εξετάσουμε το κατά πόσο υπάρχει παράβαση τέτοιου είδους κανονισμού. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη ότι μπορεί να επανέλθουμε γύρω στις 9 το βράδυ. Επομένως, παίρνουμε τη νομική συμβουλή και θα πράξουμε πάντοτε βάσει των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποσύρουμε το αίτημα και αποχωρούμε, θα διαβολευτούμε και θα επανέλθουμε στις 9 απόψε το βράδυ. Πρόεδρο. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βούλφ, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Κοιτάξτε, εγώ διέκοψα, μάλλον διέκοψα τη συνεδρίαση για κάποιο χρονικό διάστημα γιατί επικρατούσε χάος στην αίθουσα. Και ως εκ τούτου ε, εκμεταλλεύτηκα μία από τις προνομίες μου και έλαβα αυτή την απόφαση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχει την καλοσύνη, αναφέρομαι στο άρθρο 22 και θα ήθελα να σας παρακαλέσω επίσης στην Ολομέλεια να μην κάνετε τηλεφωνήματα, να ακούτε τι λέει η Πρόεδρος, γιατί τελειώς δεν θα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, όσοι θα προχωρήσουμε στην ψηφορία. Όσοι θέλουν να σταματήσει η συζήτηση θα ψηφίσουν όχι. Όσοι θέλουμε να συνεχίσουμε θα ψηφίσουν ναι. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Mindenki követhet el hibát, én is Όλοι μπορούν να κάνουν κάποιο λάθος και εγώ έκανα λάθος. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στις ε, συγκεκριμένες ε, συνθήκες και θα ήθελα παρακαλώ να δείξετε κάποια κατανόηση. Δηλαδή δεν εξήγησα με απόλυτη σαφήνεια τι σημαίνει το ναι και τι σημαίνει το όχι. Μιλάμε για διακοπή συνεδρίασης, άρα δηλαδή η ψηφοφορία είναι το αντίθετο από αυτά που είχα πει προηγουμένως. Ελπίζω να το χαίρεστε αυτό και ελπίζω και να χαμογελάτε γι' αυτό. Ξέρετε όμως, ε, αν κάποιος κάνει λάθος, ε, είναι να το παραδέχεται το λάθος. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψηφίσαμε λοιπόν. Η συζήτηση λοιπόν θα συνεχιστεί από ό,τι βλέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι, από τις 9 ε, η ώρα που είπατε και μετά το βράδυ ότι θα επανέλθετε πάλι με το ίδιο αίτημα, δεν θα σας το επιτρέψω. Τελειώσαμε λοιπόν για τώρα και δίνω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια που είναι η κυρία Βαλεντσιάνο για τρία λεπτά. Θέλετε εσείς να μιλήσετε επί διαδικαστικού. Κύριε Βαλεντσιάνο, έχει το λόγο.